Λοιπόν, χαίρετε. Να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Επίτροπο Κατάινεν, στην Επιτροπή ΕΜΒΗ για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ που συστηματικά δεχόσαστε τα αιτήματά μας για ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία ε, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας στείλει σημαντικό νομοθετικό έργο ή που επεξεργαζόμαστε. Ό,τι θα αναφέρετε λοιπόν σήμερα ούτως ή άλλως είναι ε, μεταξύ των προτεραιοτήτων μας. Ε, δεν ξέρω αν ε, συντονίζεστε Ε, μόλις ε, ήμουνα και από τα, στα θέματα ευρωπαϊκής υγείας, δεν ξέρω αν συντονίζεστε και σε αυτά και αν θα αναφέρετε κάτι. Ε, το πιστοποιητικό συμπληρωματικής προστασίας, το οποίο θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική καινοτομία στο φαρμακευτικό τομέα. Βεβαίως γνωρίζω ότι κυρίως σας ενδιαφέρει η κυκλική οικονομία και τα χημικά. Να σας δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως και από εκεί και πέρα ε, θα γίνει μια ανταλλαγή απόψε με τους αδέλφους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πάντα καλό να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Αυτή τη φορά θα ε, σταθώ στην ε, αρχική μου παρέμβαση στην κυκλική οικονομία, αλλά όπως ξέρετε μας ενδιαφέρει και το θέμα του πιστοποιητικού και τα θέματα προστασίας, αν χρειαστεί. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, θα προσπαθήσω. Όπως γνωρίζετε, ε, έχουμε προχωρήσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Το 80% των δράσεων έχουν ήδη παρουσιαστεί ή εγκριθεί οι προηγούμενες δράσεις μας ε, και οι δέσμοι μέτρων που εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο θα ενισχύσουν θετικά ε, τα διάφορα βήματα για την ε, ανακατεύθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας προς μια κυκλική οικονομία. Η δέσμη μέτρων έχει τέσσερις συνιστώσεις. Η πρώτη είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά, ε, πλαίσιο παρακολούθησης δικτών, τρίτον διεπαφή μεταξύ χημικών προϊόντων και ε, νομοθεσίες περί και, ε, αποβλήτων συγγνώμη, και τέταρτον πρώτες ύλες. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τη στρατηγική για τα πλαστικά. Η στρατηγική αυτή αντιπροσωπεύει ε, ένα πολύ καλό λόγο για ε, καινοτόμα πλαστικά τα οποία ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται και ε, πάλι στην παραγωγή και αυτό δημιουργεί θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική προσπαθεί να ε, υποχρεώσει σε αλλαγέ με συγκεκριμένες δράσεις. Καταρχάς, ε, βελτιώνοντας ε, τα οικονομικά και την ποιότητα των πλαστικών και την ανακύκλωση. Μέχρι το 2030 όλες οι πλαστικές συσκευασίες πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες και ανακυκλώσιμες. Αυτό θα γίνει μέσω καλύτερου σχεδιασμού και με προώθηση ανακυκλώμενων υλικών υψηλής ποιότητας ξεκινάμε μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για να ε, προωθήσουμε τη χρήση καλών ποιοτικών πλαστικών και με άλλα λόγια, για να τα πλουστεύσω λίγο τα πράγματα, θέλουμε να έχουμε μια ενιαία αγορά για την ανακύκλωση των πλαστικών. Δεύτερον, ε, πλαστικά απορρίμματα ε, και μικροπλαστικά, βιοδιασπόμενα και πλαστικά μιας χρήσης ε, και ρήπανση στους ωκεανούς από πλαστικά. Όλα αυτά θα συζητηθούν και θα δούμε τη χρήση των πλαστικών, απογορύπτοντας τη χρήση των μικροπλαστικών, ιδιαίτερα σε κάποια προϊόντα και προωθώντας τα βιοδιασπόμενα πλακτικά πλαστικά. Επίσης, καινοτομία ε, στην ε, ε, αλυσίδα αξιών. Χρειάζονται περισσότερες ε, καινοτομίε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αποδείξουμε ότι υπάρχουν λύσει. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει ε, ένα θεματολόγιο καινοτόμα έρευνα για τα θέματα αυτά και μέχρι το 2020, το ορίζοντα 2020 για την έρευνα και την καινοτομία θα δώσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τι καινοτομίε για τα πλαστικά. Η ε, αύξηση τη ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά γίνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να υπάρχει χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας και στήριξη για αυτά τα θέματα. θα πρέπει να βελτιώσουμε την δανειοδότηση αυτών των προγραμμάτων ε, και να προωθήσουμε κατάλληλες επενδύσεις. Και τέταρτον, δράσεις ε, για τη ρήπανση από τα πλαστικά. Αυτό χρειάζεται όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να έχουμε μια απτή συνεργασία με τρίτε χώρες ε, για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσεις για τα πλαστικά, όπως για παράδειγμα καλύτερες πρωτοβουλίες για τα πλαστικά. Η στρατηγική για τα πλαστικά είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά επίσης και με τον κλάδο, τα κράτη-μέλη, τους χρήστες, τους καταναλωτές και την κοινωνία των πολιτών. Δύο λόγια τώρα για ε, τις λιμενικές ε, εγκαταστάσεις. Για να μειώσουμε τις διαρροές πλαστικών στο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα πρόταση για τις εγκαταστάσεις ε, ε, τους λιμένες. Θέλουμε να βελτιώσουμε ε, ουσιαστικά ε, τις εγκαταστάσεις αυτές και ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα σκάφη θα φέρνουν τα απόβλητά τους στους λιμένες και δεν θα τα απορρίπτουν στη θάλασσα. Ένα άλλο στοιχείο στη δέσμη μέτρων είναι το πλαίσιο παρακολούθησης, το οποίο αποτελείται από 10 βασικούς δείκτες που αναπτύχθηκαν για να μετρήσουμε τι πρόοδος έχει επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο ε, θα παρακολουθούμε τις βασικές τάσεις ε, προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε εάν αναλαμβάνονται επαρκείς δράσεις. Αυτό θα επιτρέψει στους ηθένοντας να βρουν τις καλύτερες πρακτικές και να δώσουν προτεραιότητες σε τομείς ε, που χρειάζεται το πλαίσιο παρακολούθησης ε, δεν είναι απλώς ε, σημαντικό για τους ηθήνοντες, ε, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται από όλους, είτε πρόκειται για καταναλωτούς, είτε για τον κλάδο. Και επίσης μαζί με την αρχή της επικουρικότητας, οποιαδήποτε άλλη δράση περιλαμβάνει και εθνική, περιφερειακή και τοπική συνιστόσα για να υπάρχει προώθηση και σε αυτά τα επίπεδα. Θα ήθελα τώρα να σταθώ στην διαπαφή μεταξύ χημικών προϊόντων και αποβλήτων. Οι παράγωγες πρώτες ύλες είναι στο επίκεντρο της κυκλικής οικονομίας και επομένως θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέσσερα προσκόμματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα με τη χρήση αυτών των παραγόγων πρώτων υλών. Ε, καταρχάς, ε, κάποιες ουσίες που μας ενδιαφέρουν στα προϊόντα και στα απόβλητα. Δεύτερον, παρουσία ουσιών που μας ενδιαφέρουν σε ανακυκλώμενο υλικό ε, και σε παράγωγα προϊόντα. Δυσκολίες εφαρμογής κάποιων κριτηρίων. Και τέταρτον, έλλειψη σαφήνεια ε, και συνέπεια ε, στην εφαρμογή τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ταξινόμηση των ουσιών και των αποβλήτων. Θέλουμε να διευρύνουμε τη συζήτηση και να έχουμε μια ευρεία συζήτηση με το Κοινοβούλιο, με τα κράτη-μέλη και του ενδιαφερομένου και να δούμε αν οι επιλογέ που έχουμε κάνει είναι οι σωστέ. Οι δράσεις αυτές ε, θα παρακολουθούνται μέχρι το τέλος του 2019 και από εκεί και πέρα θα υπάρχει και κατάλληλη πλαισίεση με αυτά στοιχεία και από εκεί και πέρα θα περάσουμε στη δράση. Μία ακόμα δράση, η οποία αποτελεί κομμάτι της μετάβασης προς την κυκλική οικονομία, είναι μία πρόταση που εγκρίναμε πρόσφατα για την αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Θα βοηθήσει και τους καταναλωτές και όλους να έχουν ε, καλύτερη αποδοτικότητα και να αποφεύγουν τις απώλειες σε νερό. Έτσι λοιπόν, με τον τρόπο αυτό θα κλείσουμε το κενό που έχουμε στον κλάδο του πόσιμου νερού. Για παράδειγμα, μεγαλύτερη διαφάνεια στους ε, κανόνες και στις προτάσεις προς τους καταναλωτές, έτσι ώστε αυτοί να εμπιστεύουμε περισσότερο το πόσιμο νερό. Και ελπίζω πως έτσι θα έχουμε μειωμένη χρήση εμφιαλωμένου νερού. Για παράδειγμα, ε, θέλουμε να δείξουμε, γιατί έχουμε μελέτες που μας οδηγούν στο ότι η χαμηλότερη κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού θα βοηθήσει την, τα νοικοκυριά στην Ευρώπη να εξοικονομούν 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και να μειώσει τη χρήση πλαστικών φιαλών και ε, ε, να έχουμε λιγότερα πλαστικά απορρίμματα. Θα ήθελα να κλείσω με τα σχέδια για τα όσα έχουμε να κάνουμε ακόμα φέτος. Η προσπάθειά μας να πετύχουμε μια κυκλική ε, οικονομία για το μέλλον της Ευρώπης χαμηλής εκπομπής άνθρακα θα συνεχίσει και το 2018 και μετά. Φέτος θα παρουσιάσουμε το πλαίσιο για την πολιτική για όλα τα προϊόντα που με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πιο συνεκτική και θα ενθαρρύνει και το κοινό και τους ε, ιδιώτες καταναλωτές να κάνουν επιλογές οι οποίες είναι υπέρ της ε, κυκλικής οικονομίας και έτσι θα αντιμετωπίσουμε και τα θαλάσσια απορρίμματα και τη διαρροή πλαστικού στο περιβάλλον. Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε και κάποια μέτρα υποκατάστασης για τα πλαστικά μιας χρήσης και θα κάνουμε κάτι και για τα εργαλεία αλίας. Προσπαθούμε εμείς να ακολουθούμε τα όσα προτείνουμε, να μην είμαστε ο δάσκαλος που δίδασκε και λόγια δεν είναι κράτη και γι' αυτό έχουμε τη δική μας στρατηγική για τα πλαστικά, την οποία θα σεβαστούμε για να μειώσουμε τη χρήση πλαστικών θυαλών ε, και ε, στις δικές μας υπηρεσίες. Και θα δείτε τα αποτελέσματα αν μας επισκεφθείτε, οπότε θα ήθελα να προκαλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας ανταγωνιστεί σε αυτά, να δούμε ποιο από τα δύο όργανα θα είναι τελικά πιο κυκλικό σε επίπεδο εσωτερικής κατανάλωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ένα πρώτο γύρο σχολείων. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων θα του απαντήσετε και μετά θα κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς κύριε Αντιπρόεδρε Νομίζω πως το τελευταίο που είπατε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε οπωσδήποτε, γιατί ξέρετε πως ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον σε επίπεδο κυκλικής οικονομίας, ε, με πως οι στόχοι και τα σχέδια θα πρέπει να μεταφραστούν από λόγω μορφή νομοθετήματος. Και για το θέμα της υγείας είστε αντιπρόεδρος και έχουμε ανταλλάξει απόψεις για το θέμα αυτό, αλλά ξέρω, ε, νομίζω πως και τα όσα είπε ο Επίτροπος κύριος Αντριοκάητης σήμερα το πρωί ε, οδήγησαν στον αισθάνομαι όλο και περισσότερη απογοήτευση γιατί ε, σε κάποια συμπεράσματα νομίζω ότι θα πρέπει ήδη να ξεκινήσετε εσείς με την επιπτωσιολογική μελέτη με συγκεκριμένες προτάσεις που καλωθορίζω και χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα αυτή ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή των σχεδίων που έχετε για την κυκλική οικονομία. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα εκ των όνου κάνευ για όλε αυτέ τις πρωτοβουλίε και για την εφαρμογή των όσων μα προτείνεται στα πλαίσια του σχοδίου και αυτό είναι να γίνουν όλα αυτά στα πλαίσια ενό σφαιρικού πλαισίου που θα πρέπει να είναι η στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον. Χρησιμοποιώ την ευκαιρία λοιπόν για να σα ρωτήσω αυτή τη στρατηγική πότε θα την παρουσιάσετε, ποιε θα είναι οι προτεραιότητες και με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως οι πρωτοβουλίε για την κυκλική οικονομία θα ενταχθούν στα πλαίσια αυτού του πλαισίου και της στρατηγικής χωρίς να έχουμε ε, αντιφατικές προτάσεις. Είναι μια πρωτοβουλία ε, ε επίσης για την ανακύκλωση έτσι ώστε ε, αντιφατικές προτάσεις. Είναι μια πρωτοβουλία ε, ε, επίσης για την ανακύκλωση έτσι ώστε κλωμένα προϊόντα να μπορούν να χρησιμοποιούνται εκ νέου ως υλικό ε, χρήσιμο ε, και μη τοξικό. Θα ήθελα να καλωσορίσω τη συμπερίληψη των νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας ρωτώ πώς έχουμε προχωρήσει, ποιες ήταν οι προτεραιότητες, Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. γιατί η παρουσίαση που μας κάνατε ήταν πολύ σωστή και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί από κοινού μια τεράστια πρόκληση. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω το εξή. Εδώ και χρόνια έχουμε ε, νερά που ταιριάζουν με τους προέδρους μας. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί τα μπουκαλάκια με το νερό που έχουμε μπροστά μας όλοι είναι πια ιταλικά. Άρα λοιπόν, τι γίνεται με το βουνό πλαστικού που ε, μαζεύεται κάθε μέρα, ε, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και επίσης έχουμε το σχέδιο δράσης για την κυκλική ε, οικονομία που ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια και μας είπατε ότι οι ρυθμοί εφαρμογής είναι ικανοποιητικοί. Και η αλήθεια είναι πως προχωράμε. Έχουμε το πακέτο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο μήνα εκκρεμωτήτων που είναι τεράστιος πριν καταφέρουμε να πιστέψουμε ότι πετύχαμε την κυκλική οικονομία. Και έχω πολλές αμφιβολίες και αρκετές ερωτήσεις γιατί θεωρώ πως θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια καλύτερη ισορροπία πριν ε, πετύχουμε την κυκλική οικονομία. Τι γίνεται με τον οικολογικό σχεδιασμό, το eco-design, τι έχετε κάνει εσείς εκεί. Και θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία, μία προσέγγιση προς την κατανάλωση που είναι πραγματικά κυκλική και να δούμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Κάποιοι έχουν πολύ ενδιαφέροντα project αυτή τη στιγμή στα σκαριά και πιστεύω πω αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να δρέψει τα πλεονεκτήματα αυτή τη κατάσταση προ όφελο ολόκληρη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο δράση πρέπει να σα πω πω συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρα που είναι πάρα πολλά ενδιαφέροντα για τη βιομάζα. Ε, στην αναπομπή τη οδηγία για τις ΑΠΕ βλέπουμε πω μιλάμε για, την, για τα ανακυκλωμένα ε, επαναχρησιμοποιούμενα ε, υλικά και για την χρήση ενεργειακών υλικών. Λοιπόν, τι θα γίνει με τα βασικά προϊόντα και πώς αυτά όταν ανακυκλώνονται μπορούν να μας δώσουν πηγές ενέργειας. Και τι γίνεται με το πακέτο, με τα όλα τα μέτρα για το monitoring. Τι θα κάνετε εσείς για να εφαρμόσουμε στην πράση την ε, πραγματική αξιολόγηση όλων αυτών των μέτρων. Το πλαίσιο που έχουμε θα μας επιτρέψει να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα που εγκρίναμε. Και να σας πω πως συμφωνώ απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτό είναι το πέμπτο, για την απαγόρευση πλαστικών που εισάγουμε από την Κίνα, γιατί νομίζω ότι ε, εδώ έχουμε πεδίο δράσης λαμπρό για την έρευνα και νομίζω στα πλαίσια του Horizon 2020 μπορούμε να το καταφέρουμε. Όμως, θα πρέπει να δούμε πώς τα υλικά θα χρησιμοποιούνται, θα χρησιμοποιούνται με το σωστό τρόπο και θα καταφέρουμε στα πλαίσια της πολιτικής να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Και επίσης, ποια είναι τα σχέδιά σας έτσι ώστε η κυκλική οικονομία να συνεχίσει να είναι μια προτεραιότητα και μετά το 2020. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνετε τώρα για να συνεχίσουμε να διατηρούμε το θέμα αυτό ως ύψης της προτεραιότητας. Σας άφησα λίγο ε, περισσότερο χρόνο γιατί σήμερα είστε μόνο από την ECR. Αλλά περισσότερο δεν πρόκειται για διαγωνισμό, αλλά μάλλον ποιο κάνει κύκλους γύρω από τις προκλήσεις, περί τους δηλαδή, σε οδοντόκραμες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μικροπλαστικά βρίσκονται παντού. Χρειάζεται μια πάρπουμε επίσης ότι οι χώρες μέλη για την ώρα σχεδιάζουν να καταργήσουν τα πλαστικά μέσω της εθνικό ηθικολογικά αλλά ταυτόχρονα βλέπετε ότι η αγορά κατακαιρματίζεται περισσότερο και αυτό σημαίνει ένα βήμα προς τα πίσω και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μας ωφελεί. Ε, ήμουν ε, πολύ ευχαριστημένος αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια σύμβουλη για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ που τηρήσατε και τον χρόνο σας και για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. θα περιοριστώ στα δύο λεπτά. Μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ κύριε Κατάινεν έχουμε πράγματι αυτή την ετήσια ανταλλαγή απόψεων. Θυμάμαι την περισμένη φορά είχατε κάπως ενοχληθεί διότι ε, είχατε δεχτεί πολύ κριτική και ε, είχατε πει ναι κατάλαβα όλα τα κάνω λάθος. Τώρα είμαστε πιο ικανοποιημένοι, ιδίω για τα πλαστικά και θα φανεί και από τον τρόπο που ρωτούν οι συνάδελφοί μου. Φαίνεται λοιπόν ότι κινούμεθα σωστά. Αλλά εξακολουθούμε να εξετάζουμε τον οδικό χάρτη που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι ένα από τα θέματα που είναι κάπως ασαφές ακόμη είναι σχετικό και με το eco-design. Τι σχεδιάζει η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ώστε να διευρύνει το eco-design. Γνωρίζουμε ότι το eco-design μπορεί να, είναι, να γίνει πάρα πολύ αποτελεσματικό και υπάρχουν και ευκαιρίες. Αλλά τότε δεν θα πρέπει να αρκεστεί μονάχα στην αποδοτική χρήση της ενέργειας και στη χρήση των υλικών όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τώρα μας αφήνει κάπως στα σκοτεινά πριν να αναλάβει η νέα Επιτροπή. Και για τον οδικό χάρτη τίθεται το θέμα της βιομάζας. Μας περιμένει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την οδηγία για, τα, για τις αλλά και στον οδικό χάρτη υπάρχουν και παραδείγματα της ε, βαθμιδών ε, χρήσης της βιομάζας. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν από την Επιτροπή, από εσά δηλαδή, τι μπορούμε να αναμένουμε εκεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι η βιομάζα εν τέλει είναι και ένας ε, πόρος που ε, βρίσκεται σε σπάνιδα. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο και αυτή η βαθμιδόν χρήση του, της βιομάζας μπορεί να είναι μια από αυτές ε, τις προσεγγίσεις. Ευχαριστώ λοιπόν, θα χρειαστεί να περιλάβουμε όλα αυτά και στην Επιτροπή δώσετε απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αποηθέσω και πάλι τον ε, κύριο Λίζε για δεύτερη φορά σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στα όσα σας εξήγησε σήμερα το πρωί ο Επίτροπος Κάιδης Το ζήτημα είναι σημαντικό, ως γνωρίζετε όλοι. Εάν τα φάρμακα δεν αποδίδουν καλά διότι δεν είναι αρκετά καλά είτε διότι έχουν γίνει πολύ ανθεκτικά τα μικρόβια, τότε ε, πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα πρέπει να είναι η σωστή δράση. Δεν αποκλείουμε, ξέρουμε δηλαδή αν η νομοθετική δράση είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Θα δούμε ε, πώς θα προχωρήσουμε την οδηγία. Τώρα για τον ορίζοντα 2020 θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει την προσπάθεια να εξασφαλίσει νέε καινοτομίε για την ε, εξέλιξη των αντιβιωτικών. Ερώτηση ΠΟΚ. Πότε θα καταθέσει μια πραγματική στρατηγική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί θεωρούμε ότι έχουμε τη στρατηγική του 2015 η οποία πρέπει να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα. Βρισκόμαστε τώρα στην φάση εφαρμογής. Όπως είπα και εισαγωγικά, ήδη 80% των δράσεων στο σχέδιο κυκλικής οικονομίας του 2015 έχουν ήδη μπει στα σκαριά. Κατά την άποψή μου τουλάχιστον, αυτό είναι το πρώτο μπαράζ μέτρων και η πρώτη προσπάθεια να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τι ακριβώς σημαίνει η κυκλική οικονομία, σε ποιους χώρους, ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, σε ποιους τομείς για να αλλάξει το μοντέλο της οικονομίας στην Ευρώπη. Δεν είναι και το τελευταίο, η τελευταία δέσμη μέτρων κυκλικής οικονομίας, γιατί αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει και η οικονομία παρούσα Επιτροπή δεν πρόκειται να υποβάλει νέο σχέδιο κυκλικής οικονομίας, όμως αναγκαστικά θα το πράξει η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να παραμείνει ένα από τα θέματα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως στρατηγική αλλά και ως δράση. Άλλες ερωτήσεις πριν να πω περισσότερα για την κυκλική οικονομία, για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Εργάζονται οι πραγματογνώμονες για το θέμα αυτό, ως γνωρίζετε άλλωστε, και φτάνει στο πολιτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε, σε λίγες εβδομάδες ή το πολύ σε λίγους μήνες. Ίσως φέτος να μπορέσουμε να καταθέσουμε λύση. Θέμα πάρα πολύ ε, περίπλοκο, αλλά και πολύ σημαντικό και θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η γνώση του θέματος που έχουμε είναι πράγματι επίκαιρη. Τώρα για το eco-design είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό εργαλείο. Έχει δείξει απτά αποτελέσματα, γνωρίζετε άλλωστε και εσείς καλύτερα και από μένα. Το πρώτο σύνολο μέτρων με την οδηγία eco-design και energy labeling θα εξοικονομούμε ενέργεια μέχρι το 2020 που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας της Ιταλίας. Εάν μπορέσουμε να περάσουμε και τα έξι νέα προϊόντα που ελπίζουμε να μπορέσουμε να βάλουμε στην οδηγία Eco Design, θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε περίπου το ίδιο ποσό ενέργειας που καταναλώνει ετησίως η Σουηδία. Προσθέστε λοιπόν την σουηδική κατανάλωση στην ιταλική από την ε, σκοπιά αυτή. Πολλοί λοιπόν επικρίνουν, λένε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει χέρι στις μηχανές του καφέ ή ε, ε, στα στεγνοτήρια. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η οδηγία Eco Design μπορεί να βοηθήσει να επιτευχθούν σημαντικά πράγματα. Ε, καμιά φορά τα μεγάλα ποτάμια τροφοδοτούνται από μικρά ριάκια. Για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία Eco Design, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή στην παρούσα θητεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και δεν είμαι βέβαιο. Όπω είπατε, κύριε Eckhout, θα πρέπει να διευρυνθεί και με την αποδοτική χρήση των πόρων. Είναι ας πούμε ένα μεγάλο ψάρι που αξίζει τον κόπο να κάνουμε, αξίζει, το, αξίζει η προσπάθεια να το πιάσουμε. Αλλά αυτά θα χρειαστούν κάποιο χρόνο και δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα μπορέσουμε να καταθέσουμε πρόταση πολύ σύντομα. Αν μπορούσα, αν εξαρτιόταν μόνο από μένα, θα αποφάσιζα αμέσω για τη διεύρυνση πάντα του πεδίου εφαρμογή. Κάποιο μίλησε για την κινέζικη απαγόρευση εισαγωγή πλαστικού. καινοτομίσουμε Να αλλάξουμε τον κανονισμό μα και χρειαζόμαστε βέβαια και περισσότερε τεχνολογικέ καινοτομίε. Τα χρήματά, μας, τελικά πετιώνται στις ε, χωματέρε αλλοδαπών χωρών. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε ευφιέστερου τρόπους για να αντιμετωπίσουμε. Οι μέλη αναλαμβάνουν εθνική δράση και ενδέχεται αυτό να εμποδίσει ευρωπαϊκές λύσεις. Χρειαζόμαστε Το πρόβλημα είναι τώρα ότι χρησιμοποιούνται πάρα πολλά διαφορετικά πλαστικά ως συσκευά. Είναι πλαστικά προέρχονται από ανακύκλωση. Άρα 94% είναι παρθένο πλαστικό που βγαίνει δηλαδή από το πετρέλαιο. Αυτό ορίζει την ποιότητα του πλαστικού. Δεν τη γνωρίζει τώρα εάν είναι χρησιμοποιημένο το πλαστικό αυτό, δηλαδή αν είναι ανακυκλωμένο. Πάλι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά για τα ανακυκλωμένα. Ο δήμο του Φράιμπουργκ στη Γερμανία, υπάρχει κάποιο εδώ από το Φράιμπουργκ. Ο δήμο λοιπόν του Φράιμπουργκ δίνετε ένα ευρώ και σας δίνουν ένα κύπελο από σκληρό πλαστικό και εάν μπορείτε το χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε και όπως θέλετε. Ε, μετά όμως μπορείτε να το επιστρέψετε στην καφετέρια ή στο βενζινάδικο που σας πούλησε το καφέ και παίρνετε πίσω το ευρώ σας. Ωστόσο ότι κατακαιρματίζεται η ευρωπαϊκή αγορά λόγω των διαφορετικών εθνικών ε, προσεγγίσεων και μέτρων. Τα μικροπλαστικά σε καλλιντικά και άλλα. Όχι, δεν είναι τεράστιε οι ποσότητε, αλλά δεν υπάρχει και λόγος να, να γίνει. Ήδη η βιομηχανία, ο κλάδος ε, κάνει, χρειάζεται να γίνει μια προσπάθεια όμως εκεί να συνεργαστούμε στο διεθνές επίπεδο. Και ε, η βαθμιδόν χρήση της. Δεν έχουμε τίποτα το νέο εδώ δυστυχώς. θα μπει στο θέμα του πηγές ωστόσο βιομάζας. Σε ορισμένες χώρες είναι πιο έντονο το πρόβλημα, αλλά όχι σε όλη την Ευρώπη. Ιδίως αν μιλεί κανείς για ξύλο. Αυτά, ας αρκεστώ σε αυτά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ο κύριος Φλόρενς είναι ο πρώτος ομιλητής. Yeah, Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να είχα ακούσει ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ποιοτικά πρότυπα για την ανακύκλωση. Το ζητούμε εμείς εδώ και πολύ καιρό. Εάν θέλουμε αγορά για την ανακύκλωση προϊόντων θα πρέπει να υπάρχουν πρότυπα. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε αγορά διότι οι αγοραστές δεν έχουν τη βεβαιότητα. Σημαντική όχι μόνο για την ενέργεια αλλά και για τις πρώτες ύλες. Διότι αλλιώς όλη η δουλειά που κάνουμε εδώ είναι για πέταμα. Και μια ερώτηση για τα πλαστικά. Θέλετε να παρακολουθήσετε όλη την ζωή και όλο τον κύκλο ζωής του πλαστικού, αλλά πώς μπορεί πιο απλό να δούμε και εδώ στο κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά τι γίνεται με όλες αυτές τις συσκευασίε μιας χρήσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Λάινεν. Εγώ είμαι επικεφαλή τη αντιπροσωπεία για τι σχέσει με την Κινέζικη Βουλή. Προέτου θα μπορούσα να σα είχα πει ότι οι Κινέζοι θα την κλείσουν την πόρτα. Θα μπορούσα να σας είχα πει ήδη από πέρσι, διότι είχαμε αντιληφθεί ότι προ τα εκεί πήγαιναν. Έχουμε τώρα ένα εκατομμύριο τόνους ε, απορρίμματα περισσότερα. Πόρτα. Θα μπορούσα να σας είχα πει ήδη από πέρσι, διότι είχαμε αντιληφθεί ότι προ τα εκεί πήγαιναν. Έχουμε τώρα ένα εκατομμύριο τόνου ε, απορρίμματα περισσότερα δεν νομίζω να προλάβουμε να τα βάλουμε στην ανακύκλωση και θα είναι κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο. Μήπως λοιπόν πρέπει να ψάξουμε λίγο περισσότερα πράγματα να βρούμε. Σήμερα το μεγάλο hit είναι τα πλαστικά στη συζήτηση μαζί σας. Πράγματι το θέμα είναι μέγα. Μέρος της ερώτησής μου είναι για τα πλαστικά πιο συγκεκριμένε ρυθμίσεις, πρότυπα. Βέβαια είπατε ότι θέλετε να φτιάξετε πρότυπα για την ανακύκλωση των πλαστικών. Πράγματι, πολλές επιχειρήσεις ζητούν ότι το λευκό χρώμα σε ανακυκλωμένο ε, δοχείο, πλαστικό, πλαστικό δηλαδή, δεν πουλιέται τόσο καλά στα ειδικά καταστήματα όσο άσπρο χρώμα μέσα σε κάτασπρο, δηλαδή καινούργια, ο παρθένο πλαστικό ε, ε, κουβά η συσκευασία. Η κυρία Γιατερμάκη. Ευχαριστούμε κύριε πίτροπε που ήρθατε. Πρέπει να σας πω ότι καλωσορίζω την ιδέα της ανακύκλωσης των πλαστικών, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τη χρήση υλικών που θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά, διότι αυτή τη στιγμή αυτά τα υλικά δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ε, τα πλαστικά σε τιμή. Ε, το δεύτερο αφορά τα προβλήματα που αφορούν ε, τα πλαστικά και τι γίνεται εκτός Ευρώπης. Ε, τι μορφής συνεργασία βλέπετε με τρίτες χώρες και δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στην Κίνα αλλά και άλλες τρίτες χώρες. Το κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Σκρίλεκ. Ευχαριστούμε κύριε Κατάινεν που ήρθατε εδώ. Καλωσορίζουμε το ε, δέσμι μέτρων για τα πλαστικά και την κατανάλωση και την περιττή χρήση πλαστικών. Κατά την άποψή μου πηγαίνετε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το μόνο ερώτημα είναι αν είστε αρκετά φιλόδοξοι. Τα μολύνουν και ρηπαίνουν μόνο τις τράπεζές μας, ε, τις ε, παραλίες μας, αλλά και άλλες εγκαταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, αυτό το μικρό φακελάκι τσάι, το οποίο ε, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης και δεν μας επιτρέπουν να αφαιρέσουμε τα μικροπλαστικά από τη ζωή μας. Ή αυτό το ε, μικρό γαλατάκι για τον καφέ μιας χρήσης. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, χρήσεις ε, πλαστικών που θα μπορούν στις ακτές μας άλλα προϊόντα. Πρέπει να τα δούμε αυτά και περιμένουμε και τι θα γίνει με τη μελλοντική νομοθεσία για τα πλαστικά μιας χρήσης. Ε, στοιχεία ε, διαχείρισης των ε, απορριμμάτων είναι το θέμα της φορολογίας. Διότι, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε προϊόντα ανακύκλωση, κύριε Κατάινε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελαή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Επίτροπε. Το πάρει μαζί του ή να το επιστρέψει. Υπάρχουν όμως εναλλακτικέ λύσεις και νομίζω ότι κυρίως είναι θέμα πολιτών και σεβασμού του περιβάλλοντός μας. Ε, θα ήθελε η τροφή μου. Τι κάνουμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρω ότι τα κράτη-μέλη διστάζουν. Ξέρω ότι η πλατφόρμα έχει ένα χάρτη πορεία, αλλά πλέον των τροφίμων που σχετίζονται με τις λανθασμένε ετικέτε τη συσκευασίε. Ε, εγώ δεν αντέχω πλέον ως γεωργός να διαπιστεύω Ευρωπαίοι πολίτες που δεν τρώνε και πεινούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πανιό. Κύριε Αντιπρόεδρε, κατά... ε, παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι επιβραδύνονται οι μπαταρίες των παλιών ε, iPhone από την ίδια την Apple για να πουλούν καινούργια iPhone. Το iPhone 8, ε, ηλεκτρικές συσκευές, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, να υπάρχει μία ε, επισήμανση που θα αναφέρεται στον κύκλο ζωής των προϊόντων. Δηλαδή, να γνωρίζει ο την ε, γαλλική πρωτοβουλία για το θέμα αυτό, αλλά επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορούμε να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε εσείς ε, λοιπόν κάποια σχετική πρώτη η κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κυρίως ε, στο πρώτο σκέλος, τη μεταφορά στην ε, ε, κυκλική οικονομία με στόχους υψηλότερης ανακύκλωσης και σημεία αναφορά στον οικολογικό σχεδιασμό, το eco-design, νομίζω ότι έφτασε η στιγμή για οδηγία. Ε, να πω και κάτι ακόμα. Εσείς ασχολείστε και με την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις. Πρέπει να δίνονται δυνατότητες για επενδύσεις σε υποδομές, ώστε να διευκολύνουμε και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να... Ε, θέματα που μας αποσχόλησαν ε, κατά τη διάρκεια ζωής του, ε, στρατηγικού, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Λίγα προγράμματα έχουν ε, εφαρμοστεί για την εξοικονόμηση πόρων και την κυκλική οικονομία. Ίσως μια πιθανή εξήγηση να είναι ότι η κυκλική οικονομία στη στήριξή μας. Ελπίζω όμως ε, ότι θα υποστηρίξετε κι εσείς και θα βοηθήσετε για να διαβιβάσουμε το μήνυμα του ε, παράγοντε τη κυκλικής οικονομία, όποιοι είναι, αν χρειάζονται οποιαδήποτε χρηματοδότηση κινδύνουν περισσότερο κεφάλαιο ε, που δεν μπορούν να βρουν στην αγορά ή ορισμένα. Τώρα, για τα πλαστικά μιας χρήσης. Έχουμε ήδη αυτή την περιβόητη δέσμη μέτρων ε, για τα πλαστικά μιας χρήσης που εφαρμόζεται με ένα βασίλειο. Υπάρχει ένα τέλος ε, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται για χρήση αυτών των πολύ λεπτών ε, συσκευασιών μιας χρήσης και αυτό άλλαξε και τη συμπεριφορά των ανθρώπων περισσότερο από ότι της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης. Και αυτό είναι και το ε, κατάλληλο παράδειγμα. Χωρίς να έχουμε μια νομοθεσία πάρα πολύ αυστηρή, ε, μπορούμε να έχουμε μια ευρύτερη προσέγγιση η οποία επιτρέπει στα κράτη-μέλη ε, να... Εάν καταφέρουμε λοιπόν να ενισχύσουμε και να επηρεάσουμε την συμπεριφορά των καταναλωτών και να αλλάξει ε, στάση ο καταναλωτής, αυτό είναι ο βασικός κινητήριος μοχλός ε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ε, το... Η πλαστικομίας λεπτής τρώσης θα το επεκτείνουμε και θα δούμε ποια προϊόντα μπορούμε να συμπεριλάβουμε. Πάντως, για παράδειγμα, προωθούμε τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης. Ίσως αυτά είναι τα πιο κατάλληλα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα καλαμάκια, για παράδειγμα, θάλασσα. Οπότε, ναι, είναι η κατάλληλη στιγμή και πρέπει να το κάνουμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τη χρήση αυτών των προϊόντων που πολύ συχνά βρίσκουμε στις παραλίες μας. Αλλά, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι σωστός ο κατάλογος των προϊόντων. Γιατί και δεν θα ήθελα να αναφερθώ και να κατονομάσω συγκεκριμένες χώρες Δεν είμαι προφήτης, αλλά σίγουρα είναι άλλες ασιατικές χώρες μάλλον οι υποψήφιες. Ελπίζουμε, δεν είμαι προφήτης, αλλά σίγουρα είναι άλλες ασιατικές χώρες μάλλον οι υποψήφιες. Ελπίζουμε πως θέλουμε ένα πρότυπο για τις πλαστικές συσκευασίες και να αντιμετωπίσουμε το εκ... Στη συνάδελφο κυρία Γιατεμάκη να πω το εξή. Θέση του... των υλικών που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά το πρόβλημα το εξή. Τα βιοδιασπούμενα γνώμη και να εξηγήσουμε τι σημαίνει βιοδιασπούμενο είναι βιοδασπούμενο υπό συγκεκριμένε συνθήκες. Χρειάζεται για παράδειγμα συγκεκριμένα... Οπότε θα πρέπει και αυτά να τα εξηγήσουμε ε, στους συμπολίτε μας και να καταλαβαίνουν και σε αυτό που θέλω είναι η κυκλική οικονομία και η πολιτική για τα πλαστικά να αποτελέσουν κομμάτι του υψηλού επίπεδου οικονομικού διαλόγου έχουμε την Κίνα και, και το κατά πόσο θα πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα. Το κοιτάμε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Για τα θέματα της φορολογίας των πλαστικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλαστικών αλλά και άλλων υλών. Δεν ξέρουμε ακόμα παραπάνω. Έχουμε μία πλατφόρμα που αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά και το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να μετρήσουμε από πού προέρχεται αυτή. Θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να γίνει. Θα είναι τα κράτη-μέλη που θα νομοθετήσουν και θα εφαρμόσουν, θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως υπόψη, είναι σοβαρό το πρόβλημα. Θέλουμε όμως να καταλάβουμε καλύτερα το τι συμβαίνει πριν να ξεκινήσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι είναι το ίδιο περίπου με την, ένε, την σήμανση της ενεργειακής ε, χρόνια, πέντε χρόνια και νομίζω ότι αυτό όντως θα επηρεάσει την ε, συμπεριφορά του καταναλωτή. Πρέπει να τα δούμε λοιπόν αυτά. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήσασταν όπως πάντα πολύ ενημερωτικός και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε σε αυτό το φάκελο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι το 2019 έτσι ώστε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εργασίας στους συμπολίτες μας.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 Okay, dear colleagues, if you take your seats, maybe Καθίστε, συνάδελφοι, για να ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Καλώς ορίσατε. Όπως ξέρετε, αυτή είναι η συνήθις ετήσια ανταλλαγή απόψεων με το Διευθυντή του Οργανισμού για να μας πει κάποια πράγμα, πράγματα για το πρόγραμμα εργασίας για το 2018 και το, ή το 2019. Πιο απ' όλα. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, τίνουμε βίκο σε όσα έχετε να μας πείτε για το επόμενο πρόγραμμα. Να αναφέρω απλώς ότι θα σας επισκεφθεί μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος το δεύτερο εξάμεινο του 2018 και βεβαίως μετά από την παρουσίασή σας ε, θα ζητήσω από τον κύριο Μπράντι και ε, όποιο συνάδελφο φυσικά ενδιαφέρεται και θέλει να θέσει ερωτήσεις να λάβει το λόγο. Πρώτα όμως η παρουσίασή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας πω τι κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ε, εδώ στην Επιτροπή σας. Καταρχάς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, πλαισιώσουμε τη δουλειά που κάνουμε ε, με μια τριπλή προοπτική όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα για το τι κάνουμε όχι μόνο το 2018 και το 2019 αλλά και αργότερα γιατί πρέπει να δούμε και πώς εφαρμόζονται όλα αυτά βάσει του κεκτημένου. Αλλά δεύτερον ασχολούμαστε ε, και ε, με ένα θεματολόγιο για το 2030 και συνεργαζόμαστε με εταίρους ε, στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχουν μέθοδοι υποβολής εκθέσεων όπως για παράδειγμα για τη μέτρηση της κυκλικής οικονομίας, της Ενεργειακής Ένωσης και των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Και όλα αυτά συνάδουν και με την μεταβατική προοπτική που επιλέξαμε στο πολιετές πρόγραμμα που εξετάζει ε, και ε, το 7ο πρόγραμμα πλάσιο και πώς μπορούμε να ζήσουμε με τα μέσα που μας προσφέρει ο πλανήτης. Ε, όλα αυτά τα βλέπουμε με την αναπτυσσόμενη ατζέντα πολιτικής της Βρυξέλλες για να έχουμε μια καλύτερη προοπτική για την παρακολούθηση τον έλεγχο και την ανάλυση της ατζέντα ε, με σύστημα. Και αν δείτε το οικοσύστημα και φυσικά και τα συστήματα της κοινωνίας που παρέχουν στους πολίτες την κατάλληλη ευημερία, και προσδίδουν οικονομική αξία. Επικεντρώνουμε τις δουλειά μα ε, στο ενεργειακό σύστημα που βλέπουμε σχέσει μεταξύ κλίματο και ενέργεια ε, και τι γίνεται με την ενεργειακή ένεση. Βλέπουμε το σύστημα τροφίμων και εδώ θέλουμε να υποστηρίξουμε την κοινή γεωργική πολιτική και τη μεταρρύθμισή τη. Επίσης να πω ότι πρόσφατα ασχοληθήκαμε και με μια έκθεση για το σύστημα των τροφίμων που δεν θεωρεί ότι η γεωργία είναι το μόνο στάδιο στη συστημική προσέγγιση για το πώς υποβάλλουμε εκθέσεις ε, και βλέπουμε πώς θα μπορούσε να μας ωφελήσει αυτό. Όσον αφορά το σύστημα, Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας και τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζο για να δούμε το θεματολόγιο για την ε, ε, αστική βιωσιμότητα και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε επίσης και την διακοπή της χρήσης του άνθρακα στις μεταφορές, ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά στις πολιτικές συζητήσεις. Να αναφέρω δύο πρόσφατες εκθέσεις ε, για την έκθεση για τις μεταφορές και το περιβάλλον, καθώς επίσης και την περσινή έκθεση που ήταν ε, για την βιώσιμη μετάβαση της κινητικότητας και η φετινή έκθεση επικεντρώθηκε στη ρήπανση από την αυτιλία και την αεροπορία, δύο φλέγοντα θέματα. Να πω επίσης ότι στη διαχείριση των γνώσεων που ακολουθούμε, που ε, βασίζεται σε παρακολούθηση, σε δεδομένα, δείκτες, αξιολόγηση και γνώσεις, Υπάρχει μια πολύ στενή σχέση ε, όσον αφορά την παρακολούθηση και τα δεδομένα. Υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις οι οποίες είναι ε, εγγεγραμμένες στο κεκτημένο. Συνεργαζόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τη Γενική Διεύθυνση Κλίμα και τους υποστηρίζουμε σε αυτή την προπτική και αυτό κάνουμε και με τα κράτη-μέλη είμαστε υπεύθυνοι για το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Δίκτυο ε, Πληροφοριών και Παρατήρησης που περιλαμβάνει πάνω από 70 εθνικούς οργανισμούς που συνεισφέρουν. Όσον αφορά τους δείκτες και την αξιολόγηση, κυρίως ε, εκεί ε, επικεντρώνουμε την ανάλυση και τις εκθέσεις μας και ελπίζουμε να προσφέρουμε γνώσεις. Μία πολύ σημαντική καινοτομία προφανή στη δουλειά μας είναι η ενσωμάτωση και δεδομένων που προέρχονται από το δορυφορικό πρόγραμμα Κοπέρνικους, ε, όπου είμαστε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που επικεντρώνεται στη συνιστόσα της γης, συνεργαζόμαστε με τις χώρες και χρησιμοποιούμε και τα ατμοσφαιρικά και κλιματικά δεδομένα και στοιχεία τα οποία παίρνουμε από το πρόγραμμα Κοπέρνικους δηλαδή. Αν δείτε τι κάνουμε όσον αφορά στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, ε, που νομίζω ότι είναι το ολοκληρωμένο πλαίσιο για το 2030. Είναι σαφές ότι ο στόχος προτεραιότητας 1 καλύπτει πολλά από αυτά, και αυτό είναι φυσικά το φυσικό μας κεφάλαιο. Ο δεύτερος όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των πόρων και της ε, οικονομίας χαμηλής χρήσης άνθρακα καλύπτει τους υπόλοιπους στόχους και όταν αναφερόμαστε σε πίεση και κίνδυνο για την υγεία και την εφημερία προσθέτουμε μερικούς ακόμα από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, στις δουλειές μας λοιπόν ασχολούμαστε ε, με τις περισσότερες από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης κατά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού μας θεματολογίου. Κάτι άλλο το οποίο κάνουμε είναι παρακολούθηση και η συμβολή μας ε, στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο μέσω των ετήσιων εκθέσεών μας. Και αν δείτε τους διάφορους στόχους προτεραιότητας, η πρώτη στήλη είναι οι προηγούμενες τάσεις και η τελευταία στήλη, και νομίζω ότι είναι σημαντική και αυτή η στήλη, είναι ε, οι προβλέψεις ε, για το 2020, τι προσδοκίες έχουμε για να επιτύχουμε τους στόχους του κεκτημένου. Ε, μη σας φοβήσει αυτό, δεν θα τις αναφέρω ένα προς έναν. Νομίζω ότι το ε, διάγραμμα ε, είναι προφανές. Όταν βλέπουμε το 2020 βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σαφές ε, κενό στην εφαρμογή και πόρο απέχουμε από τους στόχους για τους στόχους για το φυσικό κεφάλαιο. Εξετάζοντας τώρα μια οικονομία κυκλική και αποτελεσματική ω ως προς τους έχουμε μια πιο θετική εικόνα, αλλά βλέπουμε ε, ακόμα αρκετές κόκκινε κόκκινες και κίτρινες γραμμές ε, και επομένως ε, μας ενδιαφέρουν τα θέματα υγείας και εδώ έχουμε μόνο δύο πράσινες γραμμές και τα υπόλοιπα είναι κίτρινα και κόκκινα. Θα μπορούσα κάλλιστα να σας απαντήσω πιο διεξοδικά, αλλά αυτή είναι η συνολική εικόνα. Τώρα, να σταθώ πολύ σύντομα σε κάποια βασικά στοιχεία τα οποία μας απασχολούν υπό το πρίσμα ε, της καινοτομίας. Παραδοσιακά θεωρεί κανείς ότι ο οργανισμός απλώς εκπονεί εκθέσεις και όντως υπάρχουν αρκετές εκθέσεις και δείκτες, αλλά ε, τονίσαμε τα τελευταία χρόνια ότι ε, θέλουμε να έχουμε και μία προσέγγιση βάσει ενός χάρτη, τον οποίο θα μπορούμε να δούμε και θα βασίσουμε τις γνώσεις μας αυτών. Και μάλιστα πέρσι, τον Νοέμβριο, ξεκίνησε ο Ευρωπαϊκός Δίκτυς για την Ποιότητα του Αέρα στο Παρίσι, στη σύνοδο που έγινε εκεί. Ε, είναι μία έκθεση που έχει εκατοντάδες ε, αντίγραφα, ενώ γι' αυτό το δίκτυ για την ποιότητα του αέρα έχουμε πάνω από 19 εκατομμύρια hit, 5 εκατομμύρια ε, άτομα έχουν δει το χάρτη και έχουμε 714.000 ε, επισκέπτες. Ε, εκεί που δεν υπάρχουν τελίτσες στο χάρτη σημαίνει ότι είναι χώρες που δεν συνεισφέρουν και δεν μας δίνουν στοιχεία και επομένως δεν μπορούμε να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία μας για την ποιότητα του αέρα. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι ε, υπάρχει ε, πρόβλημα, αλλά τρία, ε, τρεις χώρες μεταξύ αυτών η Βουλγαρία και η Κύπρος άρχισαν να μας στέλνουν στοιχεία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Natura 2000 και το Σμαράγδι 2017, το δίκτυο αυτό. Και το αναφέρω το δεύτερο για να τονίσω πως είναι και πανευρωπαϊκή διάσταση των εργασιών που κάνουμε, γιατί αν θέλει κανείς να προστατεύσει μεγάλης έκτασης φυσικούς τόπους, αυτό είναι απαραίτητο. Έχουμε γύρω στους 325 επισκέπτες κάθε μέρα για τέτοιου είδους πληροφορίες, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς να πετύχει με μια παραδοσιακή ε, προσέγγιση ε, υποβολής εκθέσεων. Και αυτό το κάνουμε για να στηρίξουμε ε, την φύση στην Ευρώπη. Τώρα, για το θαλάσσιο περιβάλλον είναι προτεραιότητα για πάρα πολλούς λόγους σήμερα παντού και εδώ δίνουμε επισκόψεις τι συμβαίνει στις ε, θαλάσσιες περιοχές υποπροστασίες και έχουμε και σημεία εισόδου που σας ε, έκθεση ε, που έχουμε για το πόσιμο νερό. Αυτή είναι και σε χαρτί γιατί, ό, συγγνώμη, για, για, το, για την ποιότητα του υδάτων κολύμβησης και πρέπει να σας πω πως ε, μας ζητάνε 1,5 εκατομμύριο χάρτες ε, για να ξέρει ο κόσμος που χρόνια την αύξηση που έχουμε. Δηλαδή είχαμε γύρω στις 3 εκατομμύρια, 3,5 ε, ε, εκατομμύρια επισκέψεις κάθε χρόνο με μια αύξηση που μας έφερε στα 170 εκατομμύρια την περσινή χρονιά. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για το 2018 και το έκθεση που παρουσιάζουμε και θα συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν μία προσέγγιση που θα φασίζεται στη λύση προβλημάτων, όπου τέκουμε την παραδοσιακή προσέγγιση και προσπαθούμε να συνδέσουμε αυτό με την καινοτομία και τα επενδυτικά ε, ε, χαρτοφυλάκια επενδύσεων στην τον 21ο αιώνα και όχι που να βασίζεται στις παραδοχές του 20ου. Και για να κλείσω αυτή την έκθεση και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο θα ήθελα να τονίσω τα εξής έχουμε τρεις μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον, όχι μόνο για το 2018, αλλά και για το 2019 και μετά. Και είναι δίκαιο και σωστό να πούμε πόσο σχέδια τα υποβάλλουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βέβαια, μέσω της εκπροσώπησης που έχει εκεί, είναι η αβεβαιότητα καταρχήν των συζητήσεων που γίνονται για τις πολιετής ε, προοπτικές χρηματοδότησης, τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τον Brexit και βεβαίως την αβεβαιότητα, και το λέω αυτό, αν αυτές για εμάς. Επίσης, προσεγγίζουμε το τέλος του 7ου ε, προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Δεν ξέρουμε τι μορφή και διάρκεια θα έχει το 8ο, οπότε όλα αυτά ουσιαστικά οδηγούν σε, μια, σε ένα κύκλο στρατηγικής, χάραξη στρατηγικής καινοτομίας για την εξόρυξη δεδομένων και για τα μεταδεδομένα, για την πλήρη χρήση των πληροφοριών που προέρχονται από το Κοπέρνικους και για τις, τα γεωχωρικά δεδομένα εκεί, όπως επίσης και για τις φθηνές συσκευές που μπορούν να βοηθήσουν μέσω των συμπολιτών μας να παρακολουθούμε το τι γίνεται με το περιβάλλον και δεξιότητες, αλλά επίσης επένδυση σε διαφορετικές και στεναρές σχέσεις με τα κράτη-μέλη. Και βέβαια η προσέγγιση πρέπει να είναι κάπως διαφορετική. Καταλαβαίνω λοιπόν πως πρέπει να σας μιλήσω και για το θέμα των πόρων. Εμείς έχουμε ακολουθήσει μια ξεκάθαρη στις μόνιμες και στις αρνητικές προτεραιότητες που είναι πραγματικότητα και έχουν να κάνουν με την διεθνή ε, παρουσία που έχουμε, μείωση 10% εκεί τουλάχιστον και περιεριζόμαστε στην στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θεσμούς αυτούς ε, στην UNF τριπλή, ε, τριπλό συν, όπως επίσης την, σύμβαση, την συνθήκη για τη βιοπικιλότητα, όπως επίσης και στο θέμα με ριζικό τρόπο. Συνήθως εγώ δεν παραπονιέμαι. Η ε, δική μου δουλειά είναι να διαχειρίζει με αυτά που... Ε, κάποιος φωνάζει πως μα για μένα αυτό είναι ζωτική σημασία. Ενώ στο παρελθόν είχαμε περικοπές που ήταν εύκολες. Σήμερα ό,τι προτείνουμε να περικόψουμε υπάρχει κάποιος που εκθέσεων. Και βεβαίως θέλουμε να κάνουμε κάποιο streamlining. Αλλά έχουμε τους γεωργικούς φακέλους, έχουμε τα βιοοικονομικά, έχουμε την βιώσιμη χρηματοδότηση, τη βιώσιμη χαράσουν πολιτική, όχι μόνο στι Βρυξέλλε αλλά και στα κράτη-μέλη, θεωρώ πως είναι πάρα πολύ εργατικό το προσωπικό μα, πάρα πολύ δεσμευμένο και η αξιολόγηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, παρακαλώ κύριο Γκερμπράντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω να ευχαριστήσω τους κυρίους Σκούλος και Χένεκε για την εργασία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο που κάνουν ε, για τα νέα μέλη, του, τους καθηγητές Σλίνσκι και Νέη. Καλώς ήρθατε λοιπόν και εσείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, που είναι μια σημαντική στιγμή και ιδίω και λόγω ορισμένων ε, ε, εκ των μηνυμάτων που μας έδωσε σήμερα. Μειωθεί κατά 11%. 11% είναι πολύ. Είναι σαφώς ανώτερο από η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η δική μας δηλαδή, προσπάθησε να περιορίσει τις περικοπές του προϋπολογισμού. Ωστόσο αυτές έγιναν τελικά. Και εάν η EPA έχει επίσης περικοπές της τάξης 30-40% και οι διεθνείς δραστηριότητες είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Η EPA έχει επίσης περικοπές της τάξης 30-40% και οι διεθνείς δραστηριότητες είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Είναι μέγα κρίμα που ο δικός μας EEA χρειάζεται, αναγκάζεται και αυτός να κλείσει κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές. Ενώ υπάρχει μάλλον μεγαλύτερη ανάγκη τέτοιων δραστηριοτήτων. Βλέπετε εξάλλου πρόσθετα καθήκοντα που επιβάλλονται στον οργανισμό. Η πρωτοβουλία χρηματοοικονομικής ε, βιωσιμότητα και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα και θεμελιώδη και για αυτούς και για μας. Μία ερώτηση που έχω για τον κύριο Μπράινινγκς έχει ως εξή. Γνωρίζω ότι ο οργανισμός περιβάλλοντος κάνει όλο και συχνότερη χρήση δορυφόρων. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα Κοπέρνικος χρησιμοποιείται ε, πολύ από τον οργανισμό περιβάλλοντος έμαθα ότι ακούγεται η ιδέα να αφαιρεθεί η ευθύνη αυτή από τον EA και να ανατεθεί σε ένα οργανισμό που θα ασχολείται περισσότερο με θέματα ασφάλειας στην Ευρώπη. Αν αυτό πρόκειται να σημαίνει ότι κάποιες παρατηρήσεις όπως LULUCF, όπως ε, ποιότητα του αέρα, θέλω για αυτά να ρωτήσω τον κύριο Μπράινιξ ποια άποψη έχει για το θέμα αυτό. Θα αρκεστώ σε αυτά, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, ο οργανισμός του κάθε χρόνο. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό εκμεταλλεύεται ή ε, χρησιμοποιεί. Ε, Της αποτελεί ένα ενδεδειγμένο κριτήριο αξιολόγησης κατά πόσο δηλαδή γίνονται παραπομπές στις εκθέσεις σας κάθε φορά που αξιολογούμε την βιωσιμότητα της οικονομίας. Βεβαίως έχουμε κάποιες αποφάσεις που ελήφθησαν το 2013, αλλά έχω την αίσθηση ότι σε γεωργικές γέε και αλλού, δεν είναι και πολύ γνωστή η υπόθεση. Και ωστόσο σχετίζεται και με τη δασοκοπή. Ίσως να φτάσει και μέχρι τα 40%. Μιλούμε για την αποκαταστασή τους, για την επανακαλλιεργιά τους. για την αποκόψη του διοξιδίου του άνθρακος στον κύκλο αυτό. και την αφαίρεση από την ατμόσφαιρα του διοξιδίου του άνθρωπου. Η ερώτηση αναφέρεται στις υδατοκαλλιέργειες και το δυναμικό τους. Σχετικά εκτιμήσεις για τη Βαλτική θάλασσα δείχνουν ότι η ποσότητα της βιομάζας από μικροφύκη μπορούν να φτάσουν σε πολύ ύλη, δηλαδή πάρα πολύ ε, σημαντική και χρήσιμη. και για την αλυσίδα της βιοοικονομίας. Εξετάζετε το θέμα αυτό στις δραστηριότητες σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Διευθυντά. Εδώ βρίσκομαι. Πρώτα σας συγχαίρω για τη σημαντικότερο σας άλλωστε και για τους πολιτικούς των χωρών μελών. Είπατε κι εσείς ότι στη βάση των διαθέσιμων ή ποιότητα δεδομένων που λαμβάνετε εσείς από τις χώρες μέλη, όχι τα δεδομένα τα οποία δημιουργούν οι δικοί σας πηγές, υψηλές επιτυχίες σε, ορισμένα, σε ορισμένους τομείς που ελέγχεται, όπως τα, τις ανανόσιμες ενέργειες και την χρήση της βιομάζας για παραγωγή θερμικής ενέργειας. Βλέπετε δεδοτή ειδικά για μία συγκεκριμένη χώρα μέλος, θα βρείτε στη μετρήσεις κάποια ποσά που είναι αυτών και των μετρήσεων. Ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, πράγματι είναι σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία να σας ακούμε σε τακτική βάση, να κατανοούμε τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε, δυσχέρειες δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά δυστυχώς γνωρίζουμε καλά το δημοσιονομικό θέμα πλέον και θα χρειαστεί να ασκηθεί πίεση στις χώρες μέλη για να κατανοήσουμε. Υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη αντικτύπου που δείχνει ότι παραπάνω από 22,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εξετέφησαν το 2015 σε κινδύνους υγείας ή ε, μειωμένης υγιεινής και λόγω του πόσιμου νερού. Άρα, ερώτημα, πρόβλημα που έχει και οικονομική αλλά και περιβαλλοντική και ε, κοινωνιολογική πτυχή για να βελτιώσουμε την μοίρα των Ευρωπαίων πολιτών. Μιλώντας πάντα για το νερό και για την εκ νέου χρήση των ε, ήδη χρησιμοποιών νερών. Το 2014 είχε αντιμετωπιστεί ήδη το θέμα αυτό, είχε τεθεί τουλάχιστον το θέμα, νερών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και έχουν ε, εκ των υστέρων καθαριστεί. Βεβαίω, με τις αλλαγές του κλίματος, δυστυχώς η ξηρασία την οποία βλέπουμε να επεκτείνεται σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό χωρών μελών, το κόστος ε, της, ε, του καθαρισμού των νερών από τις τοπικές αρχές Thank you very much. και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η παρατήρηση γιατί η συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ε, πρώτων πυλών και συνήθως ο έτσι είναι κατά πόσον το greening, ε, η προσπάθεια μετριασμού των συνεπειών του κλίματος ήταν αποτελεσματικό. Ε, ε, αν οι διαπραγματεύσεις μειώσουν αυτά τα μέτρα greening και ε, είναι αντικείμενο επίθεση και πολλοί λένε ότι το greening δεν θα έπρεπε να γίνει και αυτό δεν είναι σωστό μάθημα. Ίσως χρειαζόμαστε λοιπόν καλή δουλειά και ανάλυση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο τώρα που θα ήθελε το λόγο. Α, συγγνώμη, έκλεισε το μικρόφωνο. Άλλος κανείς λοιπόν, αν όχι τότε να δώσω το λόγο στον καθηγητή Λένανη, που είναι από τους εκπροσώπους μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, να λάβει το λόγο για μερικά λεπτά. Η κυρία Λένανη, ευχαριστώ πολύ. Η περίοδος αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους πολίτες αλλά και από τον ε, ιδιωτικό κλάδο και λόγω αυτού πρέπει πραγματικά να ε, θεωρήσουμε ότι πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον και για τις μελλοντικές καινοτομίες. Ο οργανισμός κάνει πολύ σημαντική δουλειά και νομίζω ότι ε, κάνετε και εξαιρετική δουλειά σε θέματα παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων που είναι πάρα πολύ σημαντική ε, προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να αυξήσουμε τις γνώσεις στον τομέα αυτό. η παρακολούθηση και η συλλογή στοιχείων απαιτεί πολλούς πόρους και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι, γιατί υπάρχουν αρκετοί εταίροι που ζητούν αύξηση στη συλλογή δεδομένων. Θα ήθελα να ξέρω όμως σε ποιο βαθμό ο οργανισμός θα έχει χρόνο για να εξετάσει τη συνέχεια της παρακολούθησης των δεδομένων και να περάσει στους δείκτες, ε, στην αξιολόγησή τους και τη δράση, διότι αυτό θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό με την παρακολούθηση των δεδομένων για το μέλλον. Και ε, Σήμερα, Χάνς, μας είπατε ότι στο μέλλον θα επικεντρωθείτε στη διακυβέρνηση και στη συγκεκριμένη προσέγγιση για τα ε, διάφορες μεταβάσεις που πρέπει να γίνουν. Σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει αυτό με τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας και πώς ε, θα θέλατε να τα προχωρήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Γιάννου Λίνσκι τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε Διευθυντά. Καταρχάς, ε, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση εδώ στη συνεδρίαση και να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε για να ε, είμαστε στην υπηρεσία των εκπροσώπων σας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Μόλις ξεκίνησε η θητεία μας τις περασμένες εβδομάδες, Απλώς λοιπόν θα ήθελα επί τη ευκαιρία να σας ε, διαβεβαιώσω ότι παρακολουθώ ε, το έργο του οργανισμού εδώ και 20 χρόνια πολύ προσεκτικά και ε, έχω ιδιαίτερη εκτίμηση στον οργανισμό και αυτή τη στιγμή ε, μπορώ να δώσω μόνο συγχαρητήρια για τα προηγούμενα και τα τωρινά επιτεύγματα του οργανισμού. Τώρα, για τον υπόλοιπο κόσμο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο του οργανισμού περιβάλλοντος αποτελεί τον δείκτη της βιωσιμότητας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θεματολόγιο και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Και ε, αυτό μπορώ να σας πω ε, ότι όντως ισχύει διότι συμμετείχα στους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και γνωρίζω και τις διαδικασίες τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για το μέλλον ε, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελέσουν και ένα από τα εμπλωματικά στοιχεία υπό τα οποία θα εργαστεί ο Οργανισμός Περιβάλλοντος και βάση των οποίων θα γνωμοδοτεί προσβλέπω στη συνεργασία στην υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και θέλω φυσικά να βοηθήσω και το έργο του οργανισμού. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επιτυχία της μετάβασης και της ε, αλλαγής προς τη βιωσιμότητα ε, για να έχουμε πραγματική χρήση των φυσικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βασίζεται στην στήριξη που μπορεί να λάβει από τον Οργανισμό ε, Περιβάλλοντος της Ένωσης. Και αυτό βέβαια βασίζεται και στη στήριξη που θα λάβει από εσά, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη σας και ε, υποσχόμαστε να ε, σας υπηρετήσουμε όπως πρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι εδώ κάποιο από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και επιθυμεί να λάβει το λόγο. Όχι. Περνάμε λοιπόν. Και σίγουρα θα τα μεταφέρω και στους υπαλλήλους μας. Θα απαντήσω με τη σειρά που έγιναν οι ερωτήσεις για το Κοπέρνικους. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος και να σας πω πως σε αυτό τον κύκλο ο οργανισμός έχει νήσο πως η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του προϋπολογισμού χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη στα κράτη-μέλη και μέσω των επιστημονικών ιδρυμάτων που θα παραδώσουν δεδομένα Κοπέρνικου στα κράτη-μέλη. Έχουμε μας στο να καλύψουμε την περίοδο 2020-2027. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον οργανισμό γιατί θέλουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα μετά από τα 10 χρόνια επενδύσεων και έχουμε και το δίκτυο με τα κράτη-μέλη που θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε στο ΕΠΑ. Παρακολουθούμε το περιβάλλον, θα μπορούσε να μειώσει το βάρος για τα κράτη-μέλη και να δώσει ένα σύστημα πολύ πιο αυτοματοποιημένο. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτή την εξέλιξη και θα είμαι ειλικρινή. θα ήμασταν πάρα πολύ απογοητευμένοι. Η ευθύνη και η αρμοδιότητα, μια και εμείς έχουμε τουλάχιστον 10 χρόνια που επενδύουμε στο θέμα αυτό. Οπότε παρακολουθούμε στενά τη συζήτηση. Είμαστε σε επαφή με την Grow και με τους υπαλλήλου που είναι υπεύθυνοι για αυτό το θέμα, με τους εταίρους για το Κοπέρνικους, πως είναι πολύ σημαντικό και για τα κράτη-μέλη, μια και θα χρησιμοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του Κοπέρνικους. Ε, σύμφωνα βέβαια και με τα ποσοστά χρηματοδότησης που έχουν προσφέρει. Για το πόσο χρησιμεύουν οι εκθέσεις μας και το κατά πόσο αυτός θα ήταν ο σωστός τρόπος. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία τα πληροφοριακά τα οποία έχουμε δώσει στο Σύμβουλο ο οποίος ετοιμάζει αυτή τη μελέτη. Αυτά λοιπόν τα έχουμε θέσει στην Γενική Διεύθυνση. Θεωρούμε το Λούλου Σιέφ να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του φακέλου για το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντική αυτή η γνώση που έχουμε αποκτήσει και πολλά έγιναν στα πλαίσια του Horizon 2020. Ε, πρέπει με τους συναδέλφους στην Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα να βρούμε μια μεθοδολογία επαλήθευσης που θα ισχύσει για τη μετά το 2020 εποχή έτσι ώστε στο φάκελο αυτό να μας δώσει κάποια από τα αποτελέσματα. Πιστεύω πως αυτό αποτελεί και δοκιμή για το τι ε, καταλήγει σε στοιχεία τα οποία πολύ εύκολα μπορεί να πάρεις μέσα στο Κοπέρνικος. Για τα θαλάσσια μόλις παρουσιάσαμε ε, μία έκθεση για τα συστήματα ε, που βασίζονται ε, βάλλον. Μπορώ να σας δώσω και πιο συγκεκριμένα στοιχεία, δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά ε, και αυτό είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολούν. Για την ποιότητα των δεδομένων, για τα κράτη-μέλη και για τα δεδομένα που προέρχονται από τα κράτη-μέλη και πώς αντιμετωπίζουμε την αξιοπιστία αυτών, έχω δέωσης που είναι αυτοματοποιημένα μέσω αλγο, ε, αλγοριθμών που χρησιμοποιούνται ε, για να μας δηλώσουν ε, μέσω μηνύματος πως κάτι δεν είναι πιθανό να συμβεί ή κάτι είναι αναλυθές και έχουμε βέβαια και τους βάση αναλύουμε ε, τις βασικές ροές πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από τα κράτη-μέλη και κάνουμε μια κατάταξη με ένα σύστημα βαθμολόγησης που συμπεριλαμβάνει η χρονική στιγμή, ποιότητα των δεδομένων, συμμόρφωση με τα κριτήρια και όλα αυτά τα αναφορά που για οποιοδήποτε θέμα είναι της αρμοδιότητας μας και για το οποίο περιμένουμε δεδομένα από τα κράτη-μέλη. Είμαστε σε επαφή με τα βασικά Ινστιτούτα στα κράτη-μέλη και αν κάποια από αυτά τα δεδομένα είναι στατιστική, ε, στατιστικά δεδομένα είμαστε σε στενή συνεργασία με τα σχετικά τμήματα στη Eurostat που ασχολούνται. Να έχετε πιο λεπτομερείς ερωτήσεις μπορώ να σας δώσω και άλλες λεπτομέρειες. Πάντως έχουμε ένα πολύ σοβαρό σύστημα ε, ποιότητας, εξασφάλισης ποιότητας και ε, ε, παλήθευσης ποιότητας στις ροές δεδομένων που, ροές δεδομένων που έρχονται από τα κράτη-μέλη. Τώρα, ο φάκελος για το νερό. Είναι σημαντικό και καταλήγουμε στο ότι πάνω από 20 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν υπό συνθήκες ε, όπου το νερό ε, επηρεάζει την υγεία τους. Και εδώ το μήνυμα είναι πλήρης εφαρμογή των κανόνων, όχι μόνο στις οδηγίες για την ποιότητα του νερού, αλλά και εφαρμογή των οδηγιών για τη βιομηχανική ρήπανση και άλλου είδους ρήπανσης που τελικά ρηπαίνουν τα ύδατα. Νομίζω ότι εδώ πολλά μπορούμε να κάνουμε σε πολλά σημεία της Ευρώπης. Για το, την οδηγία για το πόσιμο νερό ε, κάνουμε πολλά. Επίσης για την... Ε, επαναχρήση του νερού ε, έχουμε κάνει και την ανακύκλωση του νερού έχουμε κάνει διάφορες ε, εκθέσεις και ασχολούμαστε με το θέμα αυτό όπως επίσης και για την επεξεργασία και βλέπουμε την αλλαγή του κλίματος, την ξηρασία. Κάναμε μία έκθεση για την επίπτωση αυτών και τις, τα τροτά σημεία ε, για μηχανισμούς απόκρισης και αντιμετώπισης και όλα αυτά όσοι έχουμε ε, και τι θα γίνει στην περίοδο της Μεσογείου αν κάποιοι θεωρούν πως οι εποχιακές, οι εποχικές ξηρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σοβαρές διαβάστε την έκθεση γιατί θα δείτε πως το θέμα θα γιγαντωθεί στο μέλλον και αν δείτε ποιες είναι οι προβλέψεις για τη ροή υδάτων ε, ε νερό πρόβλημα και για τον τουρισμό και για την γεωργία και για την στέγη οι δύο εκθέσεις που προετοιμάσαμε θα σας σταλούν. Να είστε σίγουροι. Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Κύριε Έρκη, για τους ε, μεγάλους εμπλεκόμενους στα θέματα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και για τη μελλοντική ΚΑΠ, ήμουν ένας από αυτούς που πήρε το λόγο και έκανα και μια εισαγωγική παρουσίαση. Ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε είναι εξής. Πώς μπορεί κανείς να σκεφτεί το μέλλον της ΚΑΠ και του, της αλυσίδας τροφίμων στα πλαίσια. Οποιαδήποτε πολιτική ρυθμίζει ή οδηγεί τη γεωργία με τρόπο που είναι αντίθετος με αυτούς τους ευρύτερους στόχους, που είναι στόχοι όχι μόνο ευρωπαϊκοί, αλλά και στα πλαίσια των διεθνών μας υποχρεώσεων, είναι μια πολιτική προς τη λάθος κατεύθυνση. Και θα γεωργίας των τροφίμων εστιάζουν πάρα πολύ στο γεωργικό κομμάτι αυτών, και εκεί πάει ένα μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης και παράλληλα χρησιμοποιούμε και δημόσια κονδύλια για τις αρνητικές συνέπειες αυτού του συστήματος παραγωγής τροφίμων που είναι στην υγεία μας, για παράδειγμα, τη ε, της εισόδου, ε, δηλαδή μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε τρόφιμα και μετά α, τρόφιμα στα ράφια και μετά το γεγονός ότι έχουμε τεράστια σπατάλη σε τρόφιμα ε, ίσως είναι μια καλύτερη και πρέπει να σας πω πως έχει μειωθεί το ε, προσωπικό μας αλλά έχουμε προσθέσει κάποιον για τους ε, αγροπεριβαλλοντολογικούς δείκτες και είμαστε σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για το θέμα αυτό και για τα LULUCF θα κάνουμε κάποια προσπάθεια στο μέλλον για να τα συμπεριλάβουμε και αυτά. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη μας προτεραιότητα και πρέπει να σας πω ότι γενικά με μεγάλη προσδοκία περιμένουμε να δούμε ποιον. Και αν δει κανεί το ιστορικό και το κουρίκουλουμ των δύο νέων εμπειρογνωμόνων, δεύτερο κομμάτι του τίτλου του προγράμματος εργασίας που έχουμε, η βιωσιμότητα και η μεταβατική βιωσιμότητα, ξεκινάμε από την παραδοχή. Εμείς ασχολούμαστε με ολόκληρη την αλυσίδα και θα το κάνουμε και στο μέλλον και με μεγάλη χαρά θα συνεργαστούμε και μαζί σας που είστε εμπειροί. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και πάλι κύριε Διευθυντά. του άνθρακος από, την διεθνή, ε, από τις διεθνείς αεροπορικές συγκοινωνίες. Ας αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση. Με μεγάλη χαρά ε, λαμβάνουμε την ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψη μαζί σας για το θέμα αυτό. Αυτή η απόψη εντάσσεται στο πνεύμα της τελικής συμφωνίας και είναι δεδομένη η προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Standard and Recommended Practices καθώς και για τα στοιχεία εφαρμογής. Πρόκειται για ένα ευρύ πακέτο που συναπαρτίζεται από διάφορα στοιχεία και αυτά θα σας εξηγήσει ο παρακαθήμενός μου Πίτερ. Αυτά ε, βρίσκονται σε διαπραγμάτευση και θα πρέπει να εγκριθούν στο επόμενο Συμβούλιο της ΙΚΑΟ τον Ιούνιο. Και ε, από αυτά ε, προκύπτουν ορισμένα σημαντικά στοιχεία για την θέση σε εφαρμογή της Κόρσια. Θα επανέλθουμε βέβαια μετά τον Ιούνιο διότι πρόκειται για εργασία που βρίσκεται ακόμη στα σκαριά. Πάντως, είναι χρήσιμη η παρούσα ευκαιρία να εξηγήσουμε και να σας ενημερώσουμε σχετικά με το που βρισκόμαστε. Υπάρχει νέα ε, θέση της Ένωσης Ρωμαλαίους, κανόνες εφαρμογής καθώς και συστήματα διαχείρισης που να ε, είναι αποτελεσματικά και αξιόπιστα και γνωρίζετε και εμείς έχουμε βεβαίως ε, σχετική εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πτυχές του προγράμματος αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του λογικών καυσίμων και ούτω καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ε, πρόθεσε τα θέματα αυτά, ιδίω στο Μοντρεάλ, όπως θα εξηγήσει σίγουρα πάλι ο παρακαθήμενος μου Πίτερ. Βέβαια τα πράγματα αυτά αλλάζουν. Όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία ε, θα αξιολογηθούν Θα ήθελα μάλλον τώρα να αρκεστώ σε αυτά σε ό,τι με αφορά, να υπενθυμίσω ότι πρόκειται πράγματι για κρίσιμο σημείο καμπής. Σημαντική περίοδος τώρα πριν από το Συμβούλιο της ΕΚΑΟ τον ε, Ιούνιο. Και τώρα από τη Γενική Διεύθυνση Move, ο εκπρόσωπος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ έστειλε ένα σχέδιο πακέτου Κορσία προς τα κράτη για σχόλια. Τα σχόλια πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 5 Μαρτίου του 2018. Οι ευρωπαϊκές χώρες θα διευκρινίσουν ότι αποδέχονται τη δέσμη, διότι το κείμενο ούτως ή άλλως είναι καρπός ε, μακράς και δύσκολης διαπραγμάτευσης και η Ευρώπη είναι απομονωμένη σε αρκετά θέματα. Η ευρωπαϊκή θέση εξακολουθεί ε, να είναι, όπως είπε και η συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Κλίμα, ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε εύρος τους κανόνες και διακυβέρνηση, ώστε το πακέτο κατόπιν αιτήματος από άλλες χώρες, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να κάνει σχόλια ότι θα ήθελα να ληφθούν υπόψη τα σχόλιά τους ε, σε περίπτωση που ξανανοίξει το πακέτο. Τονίζω ότι δεν θέλουμε να ξανανοίξουν εμεί οι διαπραγματεύσεις, ε, αλλά υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσουν συντονισμού σε αρκετά μεγάλο βαθμό μεταξύ κρατών μελών. Ο στόχος είναι για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ε, στην ICAG, ε, την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής αεροπορία, να γίνουν πολύ συγκεκριμένα σχόλια. Θα επικεντρωθούν στην περιβαλλοντική ακαιρεότητα του κορνία. Ε, είναι αποδεκτό βεβαίως ότι πολλά κράτη θα κάνουν σχόλια για τη δέσμη μέτρων Κορσία, ε, ο κλάδος και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις επίσης. Η διαδικασία πέραν της υποβολής των σχολείων είναι να υπάρχει ενημέρωση του Συμβουλίου της ΑΕΚΑΟ από τη Γραμματεία για τα σχόλια. Αυτό θα γίνει στις 13 Μαρτίου. Η Γραμματεία θα εξετάσει τα σχόλια που έλαβε, θα τα συνοψίσει και ε, θα δει τις συστάσεις και τα κράτη θα συζητήσουν στην Επιτροπή, ε, στην Συμβουλευτική Ομάδα της Κορσία το Μάιο και τον Ιούνιο και το Συμβούλιο του ΑΙΚΑΟ θα συναντηθεί από τις 11 Ιουνίου και για τρεις εβδομάδες. Ε, στη διάρκεια της Συνόδου του Συμβουλίου θα εγκριθούν τα όσα προτείνονται, να πω ότι υπάρχουν 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύν η Τουρκία, στο Συμβούλιο του ΟΙΚΑΟ, που αποτελείται από 36 χώρες συνολικά. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία θα έχει 8 ψήφους και θα πρέπει να προσπαθήσει βεβαίως να πείσει και άλλες χώρες, αλλά αν χρειαστεί το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Ε, εάν εγκριθεί το πακέτο Κορσία από το Συμβούλιο τον Ιούνιο, θα σταλεί και πάλι στις χώρες για να αποδεχθούν ή να απορρίψουν ε, τα πρότυπα που προτείνονται ε, στο Κορσία. Και από εκεί και πέρα οι χώρες μπορεί να επιλέξουν να υποβάλουν και τις αντιρρήσεις τους. Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία που αφορά την έγκριση αυτών των συστάσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε 73 χώρες οι οποίες αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΑΙΚΑΟ ότι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην κορσία ευθύς εξ αρχής. Ε, η Ναμίμπια, η Μποτσουάνα και η Τζαμέκα είναι οι πιο πρόσφατες προσθήκες. Εγώ λοιπόν και οι συνάδελφοί μου είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε τυχόν ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ήδη δύο άτομα που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Λίζε καταρχάς. Ο Εβραίος Συνασπισμού στην Γερμανία προβλήθηκε απέτηση να καταργηθεί το τέλος για τις, ε, από την ε, καλυπτόμενη απόσταση. Συζητούμε εδώ συχνά στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουμε μια λύση παγκόσμιου χαρακτήρα. Ε, πράγματι, δεν έχει νόημα να γίνει σε εθνικό επίπεδο, είναι προτιμότερο να γίνει παγκοσμίω, τουλάχιστον όμω σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο χαρακτήρα. Ε, πράγματι, δεν έχει νόημα να γίνει σε εθνικό επίπεδο, είναι προτιμότερο να γίνει παγκοσμίω, τουλάχιστον όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποιοι λοιπόν ευφύς άνθρωποι κάθισαν και σκέφτηκαν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της εφαρμογής του Κόρσια και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτού του τέλους που πληρώνουν ε, οι Γερμανοί επιβάτες των αεροπορικών γραμμών. Και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Κόρσια δεν έχει μεγάλη αξία. Δεν γίνονται πολλά που να ωφελούν πράγματι το περιβάλλον ή που τέλος πάντων με κάποιο τρόπο δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων μεταφορών. Το ευρωπαϊκό ETS είναι ήδη καλύτερο. Αλλά ούτε και αυτό επαρκεί ώστε να καταστήσει τελικώ περί τα, τα λαμβανόμενα μέτρα. Νομίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική διαπίστωση για όλους εκείνους που επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικοί, ε, με ίσους όρους ανταγωνισμού, η αεροπορική ε, συγκοινωνία. Διότι μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει επαρκείς προσπάθειες για να αποφευθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού τουλάχιστον στο παρελθόν. Κάναμε μια προσπάθεια με το GTS, τώρα θα αυξηθούν οι τιμές, θα έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτό, αυτή η αύξηση των ειστηρίων δηλαδή. Έχουμε δώσει εντολή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει το ποσό των δημοπρασιών του ETS θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που δεν θα έχουμε ανάγκη πλέον από εθνικά μέτρα. Ο Κόρσια ή το Κόρσια δεν είναι πάντως ο σωστός δρόμος προς την κατεύθυνση αυτή. Και αν τα αποτελέσματα του Κόρσια είναι τα προβλεπόμενα, δεν έχει κανένα νόημα να ονειρευόμαστε ότι δήθεν θα μπορέσουμε να καταργήσουμε το ευρωπαϊκό ETS για τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Συζητείτε τώρα το εάν στα πλαίσια των offset, των αντισταθμίσεων δηλαδή που αναγνωρίζονται για τις αεροπορικές επικοινωνίες, για συγκοινωνίες μάλλον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η δενδροφύτευση. Αντιλαμβάνονται πλέον και οι αεροπορικές εταιρείε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, διότι μπαίνουμε σε δύσβατα εδάφη εντό εισαγωγικών, διότι εν τέλει και οι ίδιοι οι πελάτες και οι επενδυτές ε, λένε αν αρχίσουμε τώρα να ε, επενδύουμε και στο θέμα της δεντροφύτευση, μπαίνουμε σε πολύ δύσκολα ε, λοιπόν, να την υπολογίσουμε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΚΑΟ μας, έδωσε, μας έδειξε ένα βίντεο σε μια από τις τελευταίες κοπ τα τελευταία, σε μια από τις τελευταίες κοπ δηλαδή, παράδειγμα για τον Κόρσια και νομίζω ότι τους πελάτες ούτε και τους επενδυτές. Άκουσα πόσο δύσκολη είναι όλη η υπόθεση του Κόρσια. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βρίσκεται, ας το πω έτσι, σε αξιοζήλευτη θέση, αλλά εν τέλει και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να το πράγματι εξυπηρετεί τις ανάγκες του περιβάλλοντος. Και αυτό δικαιολογεί και... Κύριο Σάικχαουτ, ε, για κάτι που διέρευσε από το κείμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ζητά την Airbus ε, για τις προδιαγραφές της, αν μπορούν να άρουν τις κόκκινες γραμμές, ναι, ανοιχτή και διάφανη. Πήραμε στοιχεία από διαρροές του χειμένου και τώρα ακούμε τις ευρωπαϊκές θέσεις μεν, αλλά εγώ δεν έχω δει κάτι επίσημο. Και πει λοιπόν θα πρέπει να είναι λίγο πιο σαφής για το τι κάνει. Νομίζω ότι είναι σοβαρό το θέμα και το γεγονός ότι δείχνεται προτιμησιακή μεταχείριση ε, συγγνώμη, αλλά στο Συμβούλιο δίνεται η αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρώπη έχει πολύ καλή εκπροσώπηση, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι σε θέση, εκτελεστική πράξη που θα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εδώ πραγματικά περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι πάρα πολύ φιλό. τουλάχιστον αυτά που κάνουμε εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εκεί ξεκινάει μια επόμενη συζήτηση, στην οποία εμεί ω συνομοθέτε θα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και από ό,τι να μειώσουμε τι εκπομπέ του αεροπορικού τομέα, και αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή ανησυχία. Ωραία. Θέλει κανείς άλλος το λόγο μετά τον κύριο Άικχαουτ. Κύριο Λάιν. Δεν ξέρω. Διερωτώ μεθα πράγματι ποιο ρόλο έπαιξε η Airbus στη διάρκεια των και για τη διαφάνεια. Μιλούμε για έγγραφα τα οποία υποτίθεται ότι δεν θα δούμε σήμερα, δεν είναι ανοιχτής πρόσβασης ούτε θέτει άλλωστε κανένα μακροπρόθεσμο στόχο για τον τομέα. Γι' αυτό ο Πέτερ ρώτησε ποια είναι τα πρόσθετα μέτρα που μπορούμε στην περαιτέρω διάταξη του Συμβουλίου του ΙΚΑΟ. Όμως μέσω του ETS δεσμευόμεθα για τα... Thank you. Uh, Mr. Thank you if you allow... Επιτρέψτε μου να μιλήσω εξ ονόματος του συναδέλφου της Τζούλι Γκέρλινγκ, που δεν μπορεί να είναι εδώ, αλλά ήταν η συγγήτρια για την πρόσφατη αναθεώρηση της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λαμβάνει υπόψη και ε, τους διεθνείς οργανισμούς πολιτικής αεροπορίας και το Κορσία. Ε, τα μέλη να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν αυτές τις συστάσεις. Χωρίς ένα αποτελεσματικό μηχανισμό εφαρμογής υπάρχει ευρύτατη μη συμμόρφωση και πολλές ε, άνθρακα. Αυτό μπορεί να γίνει όταν λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές εκπομπές ε, του χρήστη και επίσης 28C της αναδιατύπωσης για το σύστημα εμπορίας εκπομπών εκπομπών για την αεροπορία, υπάρχουν συγκεκριμένε ε, διατάξεις που ε, συνάδουν. Ευχαριστώ και τέλος ο κύριος Γκερμπράντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσία τους εδώ. Πρώτον, πολύ δύσκολο να καταπολεμήσουμε την μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και ξέρουμε όλοι ότι ο τομέας της αεροπορίας είναι ένας ετών σοβαρά. Αυτή είναι η πρώτη γενική παρατήρηση που θα θέλω να κάνω. Το δεύτερο γενικό σχόλιο είναι ότι ο τομέας των αεροπορών που διέρευσαν, το ανέφεραν και οι συνάδελφοι προηγουμένως, δεν είναι σκανδαλώδες, ε, κάτι το οποίο αφορά όλο τον πλανήτη να μην ε, συζητάτε προσωπικά και το είπα και προηγουμένως, ε, εγώ πίστευα ότι ήταν πιο κλειστό και από εκκλησία σαϊντολογίας. Αυτή την αίσθηση εξέλαβα, ότι τα πάντα που ζητά ε, ουδέτερη ανάπτυξη ως προς το κλίμα το 2020, εκεί είχαμε μεγάλη φιλοδοξία. Αλλά μετά ότι προέκυψε το σχέδιο κειμένου που έχει κυκλοφορήσει, σε μυστικά σφραγισμένα έγγραφα ή φακέλους, παρόλα αυτά, βιοκαύσιμα. Πολύ δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρετηθεί ήδη. Έχω όμω δύο πολύ συγκεκριμένε άμωση του αρχικού ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης στο ΕΚΑΟ θα δώσει τουλάχιστον μια μάχη για να ε, ε, δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσετε. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, ε, από πιο στρατηγική πλευρά, χώρες όπως η Ρωσία και η Βραζιλία είπαν σε αυτών που θα συμμετέχουν. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου σχολιάσετε και αυτά. Γιατί επιτρέπεται ακόμα κάτι τέτοιο. Uh, Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος, για τα σχόλιά σας. Επανέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών και κάπως το ίδιο αισθάνομαι, δηλαδή ένα επαναστατικό έτσι ρεύμα ε, κυκλοφορεί στην αίθουσα. Για να ακούσουμε όμως τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μπορεί ε, να κάνει περισσότερα από ό,τι σε άλλα θέματα. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις ε, του αξιωτήμους ευρωβουλευτές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Και σίγουρα η κυρία Γκράφ θα προσθέσει και άλλα πράγματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Κλίματος. Ο Δόκτωρ Λίζε μίλησε πρώτος με ερώτηση σχετικά με τα αντισταθμίσματα offset και εάν μπορεί η δεντροφύτευση να είναι επιλέξιμο κριτήριο προκειμένου. Η προσέγγιση του ΙΚΑΟ στο Κόρσια ε, έχει ως νόημα μάλλον μια απαρίθμηση κριτηρίων που θα πρέπει να σέβονται οι διαφορές μονάδες και ένα από τα κριτήρια αυτά για παράδειγμα είναι η μονιμότητα των περικοπών, άλλο είναι το ρωμαλαίον της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των περικοπών. Η προσέγγιση του ΙΚΑΟ δεν αποκλεί κατηγορίες προγραμμάτων, project. Δεν υπάρχουν αρνητικές λίστες όπως είχαμε στην Ευρώπη που αποφασίσαμε να μην επιτρέψουμε ορισμένα αντισταθμίσματα να υπαχθούν στο ETS. Χρειάζονται κριτήρια επιλεξιμότητας για τα offset, τα οποία κριτήρια επιλεξιμότητας θα εφαρμόζονται σε όλα τα προγράμματα τα οποία δημιουργούν offset και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, το συγκεκριμένο είδος offset θα επιτρέπεται. Άρα δεν ε, απαγορεύονται forestry credit Υπάρχει όμως και πρόταση στο Κόρσια να είναι οι μειώσεις αυτές ε, διαρκείς. Και υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ των δύο αυτών. Για τον κύριο Eichhout, πρώτα πρώτα ε, βεβαίω πρόκειται για το διοξείδιο του άνθρακος, για την αλλαγή του κλίματος, και ο κύριος Eichhout μίλησε για τις επαφές τις οποίες είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Airbus και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην διάρκεια της επεξεργασίας των σχετικών προτύπων. Προφανώς ερχόμαστε σε επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και δεν τρεπόμαστε γι' αυτό και σε αυτούς περιλαμβάνεται η Airbus που είναι και ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος ε, κατασκευαστής αεροσκαφών. Ήρθαμε σε επαφή και με άλλου ε, κατασκευαστέ αεροσκαφών. Το θέμα είναι ότι πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε αποφάσεις ε, με συγκεκριμένη βάση στον ΙΚΑΟ και είναι δείγμα ευθύνη να ζητήσουμε επαφή με τα ενδιαφερόμενα κοινά μέρη, stakeholder, που γνωρίζουν τα θέματα για να ενημερώνουν την Επιτροπή, απαντώντα στον κύριο Λάινεν για το εάν ακολουθήθηκαν κάποιε οδηγίε τη Airbus. Κοιτάξτε, η Κομισιόν δεν δέχεται ε, οδηγίε από την Airbus. Ενημερώνεται. Αυτό που ε, τελικώ έχει σημασία είναι ότι θα θέλαμε να υπάρχει πλήρη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα θέλαμε βεβαίω να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια στον ΙΚΑΟ και στην ε, διαδικασία ΚΕΙΠ μέσα στον ίδιο τον ΙΚΑΟ. Και εδώ έρχομαι στο θέμα του κ. Κερμπράντη, ότι δηλαδή τίποτε δεν καθίσταται κοινό κτήμα δημόσιο. Πρώτα-πρώτα τα ΣΑΠΣ για το Κόρσια. Ε, αυτά έγιναν με επαφή μεταξύ ε, ΙΚΑΟ και χωρών. Δεν έλαβε αντίγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαπιστώνω το γεγονός ότι εμεί λάβαμε ένα αντίγραφο τελικά αλλά δεν είμαστε κράτος. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα που μας βαρύνει. Αλλά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το μειονέκτημα αυτό συντονίζοντας τα κράτη που εκπροσωπούμε στην Ευρώπη και τα οποία διαπραγματεύονται μαζί μας στο Μοντρεάλ. Μιλήσατε για κάτι το σκανδαλώδες. Θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε για την επόμενη Cape Steering Group ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με την αύξηση της διαφάνειας της διαδικασίας CAPE. Χωρίς να γνωρίζω πού θα οδηγήσει αυτό, έχουμε υποβάλει σχετικά έγγραφα και παλαιότερα για την Διευθύνουσα Επιτροπή του 2016, χωρίς αποτέλεσμα φούβουμε. αλλά ε, δεν είμαστε αυ... εμείς αυτοί που βαρινόμεθα με τις τάξεις για μη διαφάνεια και ζητούμε να είναι πιο ανοιχτό ο χαρακτήρας των συζητήσεων στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά την διαπραγματευτική στρατηγική που θίξατε κύριε Κάουτ και ορισμένοι άλλοι, επεξεργαζόμεθα τα σχόλια για το πακέτο Κόρσια, παρόλο που θα μπορούσαμε να είχαμε δεχθεί το πακέτο ως έχει. Μία λοιπόν διαπραγματική τακτική θα μπορούσε να είναι να στείλουμε μια επιστολή που να λέει ότι δεχόμαστε το πακέτο, τη δέσμη, όπως είναι. Και όταν ξανανοίγουν τα πακέτα, όσο περισσότερο συζητούνται, τόσο δυσκολότερο είναι να εξασφαλιστεί πρόσθετη περιβαλλοντική ακαιρεότητα. Πάντως, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, εμείς έχουμε συνάψει σχόλια τα οποία θα επιφέρουν τροποποιητικές διατυπώσεις στο πακέτο Κόρσια για να ενισχύσει την περιβαλλοντική του ακαιρεότητα και να περιληφθούν και άλλα δεδομένα από ε, τους ε, operators. Βέβαια, θα υπάρχουν και άλλες αντίθετες δυνάμεις στο Συμβούλιο ΙΚΑΟ που ε, δεν επιθυμούν να δουν περισσότερη διαφάνεια ή περισσότερη περιβαλλοντική ακαιρεότητα. Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και καλούμεθα ε, να ε, λειτουργήσουμε με αυτό το πρόβλημα. Ε, η στρατηγική μας είναι πάντως να προχωρούμε με ενεργό τρόπο. Είναι σχετικώς ύστερη φάση αυτή. Έχει ήδη προηγηθεί μια τριετία εντατικών συζητήσεων ξεκινώντας από την συνέλευση στην οποία τη συμμετάσχει πολύ εξημών και οι λεπτομέρειες έχουν συζητηθεί. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κάνουμε τη δέσμη πιο ισχυρή. Πρέπει να εξασφαλίσουμε θα δεν θα αποδυναμωθεί. Και ένα θέμα που έθεσε ο κύριος ε, Λάινεν για τα κριτήρια βιωσιμότητα. Αριθμός κριτηρίων αφαιρέθηκε από το σχέδιο του πακέτου μεταξύ της ε, συνεδρίαση της Διευθύνουσας Επιτροπής το Σεπτέμβριο που ήρθα και ενημέρωσα την Επιτροπή σας και το Συμβούλιο του Νοεμβρίου που ενέκρινε την εκδοχή Κόρσια που υποβλήθηκε στις χώρες μέλη για διαβούλευση. Στο μεταξύ έγινε λοιπόν η διαγραφή αυτών των κριτηρίων βιωσιμότητας και αυτό ήταν μια πρόκληση για τα τρία που παρέμειναν. Το ζήτημα είναι ότι εμείς εξασφαλίσαμε τα εναπομένοντα τρία που έχουν όλα σχέση με τα ε, οξύδια του άνθρακα και διασφαλίζουμε και τα υπόλοιπα να συζητούνται ακόμη από το ΚΕΙΠ και εξασφαλίσαμε ακόμη στην απόφαση του Συμβουλίου ότι τα άλλα αυτά κριτήρια θα επανενταχθούν στο τέλος της επόμενης φάσης μέχρι το 2023. Στο μεταξύ πολύ, πολύ μικρές ποσότητες βιολογικών καυσίμων χρησιμοποιούνται στις αεροπορικές μεταφορές. Δεν μας άρεσε αυτό που θεωρήσαμε οπισθοχώρηση τον Εύριο, αλλά συνεχίσαμε μια διαδικασία να περιληφθούν τρία σημαντικά κριτήρια που είναι αυτά τα οποία αναφέρονται σε περικοπές σε ε, μειώσεις μάλλον αερίων του θερμοκηπίου με χρήση βιολογικών καυσίμων. Μιλήσαμε και για περισσότερα κριτήρια βιωσιμότητας στο μέλλον. Τίποτε από αυτό δεν υπήρξε εύκολο. Και πολλά από αυτά που είπατε εσείς κύριε Κυπράντη, κυρίως Ρωσία, Βραζιλία, γιατί φωνάζουν τόσο πολύ όταν δεν εντάσσονται καν στο Κόρσια, θα μπουν σε αυτό εφόσον θα γίνει από το 2027 και μετά δεσμευτικό για όλους αλλά δεν εντάχθηκαν οικειοθελώς. Αλλά είναι μέλη του ΙΚΑΟ, του Συμβουλίου ΙΚΑΟ. Και δυστυχώς η ψήφος για τις διατάξεις αυτές δεν αποτελεί, δεν έχει ως προϋπόθεση την οικειοθελή συμμετοχή εξ αρχής. Έχουν λοιπόν και ψήφο και φωνή και βέβαια γνωρίζετε ότι είναι χώρες των λεγόμενων BRICS Λυπούμεθα για το γεγονό ότι δεν συμμετέχουν και αλλά δεν μπορούμε και να τι εξαναγκάσουμε. Αλλά από στρατηγική άποψη νομίζω ότι διαπραγματευόμαστε όσο πιο σκληρά μπορούμε. Και η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι είναι και πάνω από του μισού οικειοθελώ συμμετέχοντε που είπαν ότι θα χρησιμοποιήσουμε το κόρσια από την αρχή και τα προβάλλουμε αυτά ω επιχείρημα. είπαμε, είμαστε από του πρώτου και πρέπει να ακουστεί η φωνή μας και ακούγεται, αλλά δεν είμαστε και σε θέση βέβαια να επαγορεύουμε τις εκβάσεις, δυστυχώς. Για την κυρία Ντεμέρσμακερ, γιατί η μη συμμόρφωση στα ΣΑΠΣ, να σας πω πως στην περίπτωση που δεν εφαρμόζονται θα πρέπει να βρει κανείς ένα διαφορετικό σύστημα. Και αν δεν τα χρησιμοποιείτε, εσείς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα άλλα κράτη-μέλη και να λάβουν μέτρα εναντίον σας. Οπότε πιστεύω ότι εδώ υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Πάντως, αυτά είναι τα νομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και αν θέλει το ΙΚΑΟ να κάνει οτιδήποτε, τότε θα πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλο φορμάτ, δεν υπάρχει ε, κάτι άλλο. Θα έχουμε και τη συγκεκριμένη σύμβαση για το θέμα, αλλά μην ξεχνάτε πως έχουμε μία σειρά από αρκετές τους τέτοιους κανόνες που έχουν να κάνουν ε, με τα επίπεδα θορύβων, με τις εκπομπές, με ε, διοξείδιο του άνθρακα, με τα πρότυπα ασφαλείας. Οπότε δεν είναι ένα μικρό θέμα ασφάλειας, είναι κρίσιμο και γι' αυτό ε, πιστεύω ότι θα φτάσουν μέχρι εκεί, γιατί αυτό είναι ό,τι πιο ισχυρό μπορούν να κάνουν. Το ζήτημα δεν είναι ε, βέβαια αν θα τα εφαρμόσετε εσείς ή όχι, αλλά το γεγονός πως άλλα κράτη-μέλη μπορούν για παράδειγμα να σας απαγορεύσουν το να πετάτε στη χώρα τους και επιτρέπεται αυτό εάν δεν έχετε ε, ε βάλει σε ισχύ κάποιο app. Εάν το έχετε κάνει, δεν μπορούν. Οπότε, θα κλείσω λέγοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη προσπαθούν αυτή τη στιγμή σε επίπεδο η να συζητήσουν αυτά τα θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος και βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστούν. Δεν γνωρίζω την απάντηση που θα δοθεί, αλλά στα πλαίσια της Κόρσια όλα αυτά θα φανούν, θα διαπραγματευτούν και να ξέρετε πως παρακολουθούν όλοι το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξέρουν πως τουλάχιστον εμείς θα εφαρμόσουμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε, τότε προφανέστατα ε, είναι λιγότερη επιτακτική ανάγκη και των υπολείπων να τα εφαρμόσουν κατά τη στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Πίτερ. Θέλω και εγώ να συμπληρώσω για κάποια θέματα ε, τα οποία ακούστηκαν για αυτά τα credit για τα δασικά, για τη δασοκομεία. Καλό είναι να σκέφτεται κανείς σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι μορφή θα πάρει η όλη διαδικασία. Ξέρετε πως ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά είναι δύσκολα βέβαια. Ε, στον ΙΚΑΟ έχουμε ένα ε, σχέδιο κειμένου, ένα σχέδιο πακέτου, όχι στα ΣΑΠ μέσα, αλλά σε κάποια άλλη διαδικασία, κάποια γενικά, πολύ γενικά κριτήρια για την επιλεξιμότητα των μονάδων και η αλήθεια είναι πως ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα κριτήρια και τελικά αυτό θα το αποφασίσει το Συμβούλιο ΙΚΑΟ δεν είναι ακόμα ε, τόσο σαφής γιατί υπάρχει ε, και η δυνατότητα της ε, εφαρμοστικής μεταγραφής το οποίο σημαίνει ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε την απόλυτη μορφή και αυτό που ξέρουμε από τις συζητήσεις που τρέχουν είναι πως πολλοί από τους εταίρους μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ζητούν να επιτρέπεται και αυτό το credit της φύτευσης δασών. Και όλα αυτά θα είναι κομμάτι του καταλόγου των αντισταθμιστικών μέτρων που μπορούν να δοθούν. Θεωρώ λοιπόν πως τα δασικά θα παραμείνουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Και αυτό δεν θέλω να το ξεχνάτε. Εγώ μίλησα περισσότερο για τη διαδικασία, για το ποιος λαμβάνει αποφάσεις, τι θα γίνει στο τέλος και πως ε, έχουμε τη θέση του πτήσουμε στο Μόντρεάλ στην συνέλευση και το οποίο φαίνεται στο ψήφισμα είναι η διπλή μέτρηση γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το έχουμε θέσει στα πλαίσια των εφαρμοστικών ε, ζητημάτων, αλλά δεν έχει κλείσει. Βεβαίως από την οπτική του κλίματος γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι